Συνάδελφοι, επανέναρξη της Συνόδου. Έχουμε μια σειρά από ε, ανακοινώσεις. Υπάρχουν τα πρακτικά της χθεσινής συνεδρίασης. Υπάρχει κάποια παρατήρηση. Όχι. Εκ των προτέρων εγκρίνονται τα πρακτικά.